Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Καλώς ήλθατε όλοι. Κηρύττω την έναρξη της ε, συνεδρίασης της συνέλευσης των Προέδρων που αφορά την ε, παρουσίαση των ε, συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την, επόμενη, από την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Φαν Ρομπάη και τον κύριο Μπαρόσο, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Καλώς ήλθατε. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν. Καταρχήν, όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν δέχτηκε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις Ολομέλειες του Στρασβούργου. Εγώ φυσικά ως πρόεδρος θα πρέπει να υπακούσω στην ε, θέληση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα λάβω το ταχύτερο δυνατόν τα μέτρα για να υπάρξει η σωστή ε, διευθέτηση των κοινοβουλευτικών εργασιών Και φυσικά θα ήθελα να προσκαλέσω και την Κομισιόν και το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στην επόμενη αυτή συνεδρία θα γίνει και η συζήτηση και η λήψη απόφασης για το νέο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων στο Στρασβούργο. Λοιπόν, στις 10 Ιανουαρίου η συνέλευση των Προέδρων θα εξετάσει το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα τεθεί μέσα στη βδομάδα τη πρώτη αυτή ολομέλεια στο Στρασβούργο του Ιανουαρίου σε ψηφοφορία. Μπορώ λοιπόν να περάσω στο κύριο θέμα τη ε, συνέλευση των Προέδρων. Θα ήθελα καταρχήν να ρωτήσω αν έχετε κάποια διαδικαστικά θέματα ή αν έχετε αντίρρηση με την ημερήσια διάταξη, εάν όχι. Κύριε Οτή, μάλιστα. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επί του έρθου 15 της συνθήκης. Στο σημείο 6 προβλέπετε ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα κάνει μια παρουσίαση μετά από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και αναρωτιέμαι γιατί γίνεται η παρουσίαση στην διευρυμένη διάσκεψη των Προέδρων εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν κατανοώ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την έδρα μας στο Στρασβούργο. Δεν έχει κανένα θέμα να κάνει με τις δυσκολίες που έχουμε εμείς τα κτίρια στις Βρυξέλλες. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μην μετατρέπονται οι πολιτικοί θεσμοί, τα πολιτικά όργανα του Κοινοβουλίου μας σε ολομέλεια χωρίς λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ποντή. Λαμβάνουμε υπόψη την παρέμβασή σας. Το ταχύτερο δυνατόν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι ενώπιον του Κοινοβουλίου για να δώσει την έκθεσή του σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά η χρονική αλληλουχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την επόμενη συνεδρία σε ολομέλες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα γίνει από τις 14 Ιανουαρίου και μόνο ενεθάρρυνε, αν θέλετε, τις κοινοβουλευτικές ομάδες μεταξύ των οποίων και η δική σας ε, πολιτική ομάδα και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να συγκαλέσουμε την ανοιχτή σε όλου του βουλευτέ τη συνέλευση των Πρόεδρων για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου το ταχύτερο δυνατό, όχι βέβαια ενώπιον τη Ολομέλεια, αλλά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ω εκπροσωπείται από την συνέλευση των Προέδρων των πολιτικών ομάδων ανοιχτή σε όλου του βουλευτέ. Υποθέτω λοιπόν ότι αποδέχεστε αυτή τη διαδικασία η οποία μας επιτρέπει να συζητήσουμε με τον κύριο Μπαρόσο και τον κύριο Φαν Ρομπάι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πολύ πιο βραχή από ό,τι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Φαν Ρομπάι. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλή εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αξιοσημείωτη εβδομάδα. Την Δευτέρα ήμασταν στο Όσλο, μετά οι Υπουργοί Οικονομικών ε, κάλυψαν τις χρονικές ημερομηνίες που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συμφωνήσουν για τον ρυθμιστικό μηχανισμό για τις τράπεζες που θα συζητηθεί συνέχεια με το Κοινοβούλιο σας. Έχουμε θέσει ένα ακρογωνιαίο λοιπόν λίθο στο δρόμο για την Τραπεζική Ένωση. Την Πέμπτη ελήφθη μια απόφαση για την Ελλάδα, θέτοντας την Ελλάδα σε ένα δρόμο βιώσιμο για την ανάκαμψη και τονίζοντα ότι η Ευρωζώνη έχει 17 μέλη και θα συνεχίσει να έχει 17 μέλη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με την μελλοντική πορεία τη Ευρωζώνη, εστιάζοντα σε δύο κύριου τομεί όπου είναι απαραίτητα περαιτέρω βήματα πέραν αυτών που έχουν ήδη συμφωνηθεί μέχρι στιγμή. Πρώτα απ' όλα, η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος. Η πρόοδος η οποία επιτεύχθη εδώ για την διαδικασία του λεγόμενου SSM είναι μια πραγματική τομή. Με το νέο αυτό σύστημα ενισχύουμε το τραπεζικό μας σύστημα. Αν είχαμε μια τέτοια μορφή εποπτείας πριν από 10 χρόνια, η χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα ήταν τόσο οξία στην Ευρώπη. Επιτύχαμε μια συμφωνία αυτή μέσα σε λίγους μήνες τον Ιούνιο δεν υπήρχαν παρά μόνο τα ψήγματα μιας συμφωνίας. στη συνέχεια, επί τη βάση των, της έκθεσης των τεσσάρων προέδρων, ετέθη η Γενική Κατεύθυνση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κομισιόν κατέθεσε τις προτάσεις της και μέσα σε τρεις μήνες οι Υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε μια συμφωνία και τώρα το Κοινοβούλιο έχει και αυτό σταθμίσει τη θέση του σε επίπεδο επιτροπών και είναι έτοιμο να προωθήσει την ε, νομοθετική διαδικασία ως την περάτωσή της τον Ιούνιο. Ζητήσαμε από τους υπουργούς να έχουν μια συμφωνία επί των λεπτομεριών του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού SSM και το επέτυχαν. Αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να πάρει έγκαιρες και αποφασιστικές αποφάσεις και αυτό είναι η λιδία λίθος της αξιοπιστίας μας. Η συμφωνία και των 27 χωρών μελών για το μηχανισμό SSM εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία αντιμετωπίζει τι ανάγκε των χωρών τη Ευρωζώνη, αλλά παραμένει ο μηχανισμό αυτό ανοιχτό σε όλου και λαμβάνει υπόψη τι θέσει αυτών που επιλέγουν να μην συμμετάσχουν. Είναι ένα ενιαίο σύστημα εποπτεία, αλλά με μια λογική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα και των Εθνικών Εποπτικών Αρχών. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξασφαλίζει στο εσωτερικό της μια σαφή διάκριση μεταξύ εποπτικών δραστηριοτήτων και τη νομισματική πολιτική. Και επίση με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε μια ενιαία αγορά για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Δεν σταματούμε όμω τι προσπάθειέ μα εδώ. Ατενίσουμε ήδη το επόμενο ή τα επόμενα βήματα που είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον τη Ευρωζώνη. Όπω ξέρετε, όλα αυτά τα θέματα αντιμετωπιστήκανε επί τη βάση τη έκθεση που προετοίμασα εγώ μαζί με τον πρόεδρο Μπαρόσο, τον πρόεδρο Ντράγκη και τον πρόεδρο Ιούνκερ το έγγραφο αυτό εργασία βασίζεται στην ενδιάμεση έκθεση που παρουσιάστηκε το προηγούμενο Οκτώβριο και λαμβάνει υπόψη τι σημαντικέ σύμβολε τη Κομισιόν στην γενική αυτή κατεύθυνση και επίση και από την πλευρά του Κοινοβουλίου ή από την έκθεσή σα συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική τη Νομισματική Ένωση και την εποπτική διαδικασία τη Μαριάν Τίσεν. Και εγώ μίλησα με την κυρία Τάισεν και με την πρόεδρο τη Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων και Απασχόληση, την κυρία Περβόν Μπέρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να θεσπίσει στο πρώτο ήμιση του 2013 ένα λειτουργικό πλαίσιο το οποίο συμπεριλαμβάνει και τον ορισμό των ιστορικών κατά κάποιο τρόπο μέσα εισαγωγικά στοιχείων ενεργητικού, ώστε στο μέλλον ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα θα έχει τη δυνατότητα να ανακεφαλαιοποιεί άμεσα τι τράπεζε βάσει μια τακτή διαδικασία για τον μηχανισμό αυτό εποπτεία το SSM, να είναι πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό, αποφασίσαμε επί τη βάση τη εκθέσεω των τεσσάρων πρόεδρων ότι όταν λειτουργήσει αυτό ο μηχανισμό, θα πρέπει να υπάρξει και ένα ενιαίο μηχανισμό επίλυση τραπεζικών ιδρυμάτων με τι απαραίτητε εξουσίε για να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τράπεζα στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν μπορεί να επιληθεί με τα κατάλληλα εργαλεία. Κατά τη διάρκεια του 2013 η Κομισιόν θα υποβάλει μια πρόταση η οποία θα πρέπει να τύχει εξάρτηση κατά προτεραιότητα με στόχο να υπάρξει η έγκριση της πρότασης αυτής μέσα στον τωρινή κοινοβουλευτική θητεία. Ο στόχος είναι η μείωση των κινδυνών για τους φορολογουμένους και για την οικονομία με το να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε αποτυχία τράπεζας θα αντιμετωπιστεί με ταχύ και τακτικό τρόπο και τελικά θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί καταρχήν από τον ίδιο το χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό θα είναι ένα ακόμα μείζον βήμα προ τα εμπρό. Όλα αυτά με φέρνουν μετά από την πρόοδο για την Τραπεζική Ένωση σε ένα δεύτερο τομέα όπου εστιάσαμε την προσοχή μας στο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι οικονομικές πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχουν μια μεγαλύτερη σύγκληση. Το σημείο ακίνησης μας είναι απλό. Η οικονομική πολιτική είναι θέμα κοινού συμφέροντος, ζωτικού συμφέροντος για τις χώρες όλες αυτές που βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα νόμισμα και 17 διαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Κάποια από τα κράτη-μέλη μας είχαν προβλήματα ε, οικονομικής διαχείρισης για πολλά χρόνια και καθυστέρησαν πάρα πολύ να αναλάβουν δράση. Ως πρόεδρος λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω προτινόμενα μέτρα και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οδικό χάρτη που δεσμεύεται χρονικά προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013 με συνεργασία του Πρόεδρου της Κομισιόν και φυσικά μετά από μια διαδικασία διαβούλευσης. Αυτά τα τέσσερα θέματα που θέλω να παρουσιάσω είναι τα εξής. Πρώτον, συντονισμό των κυρίων των σημαντικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένε χώρε και αυτό περιλαμβάνει και διαστάσει εξάντια. Δεύτερον, την κοινωνική διάσταση τη νομισματική ένωση που περιλαμβάνει και κοινωνικό ε, διάλογο. Η, τρίτον, τα συμβόλαια ανταγωνιστικότητα μεταξύ των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέταρτον, τον μηχανισμό αλληλεγγύη, ο οποίο μπορεί να ενισχύσει τι προσπάθειε οι οποίε καταβάλλονται από τα κράτη-μέλη, τα οποία δέχονται τέτοιε συμβατικέ σχέσει, συμβόλαια δηλαδή ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά δεν αποτελούν αυτοσκοπούς. Ο γενικός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα της νομισματικής ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση σε όλη την Ευρώπη. Μπορούμε να επιβιώσουμε σε μια παγκοσμία οικονομία μονάχα εάν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και σε τελική ανάλυση εξαρτάται από την απόδοση της πραγματικής οικονομίας για να εξασφαλίσουμε μια λειτουργούσα και υγιή, οικονομία. Πολλοί το λησμονούν αυτό το θέμα. Όλοι συμφωνούμε ότι μέσα στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι συνεχίσουμε να έχουμε δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία σε ένα επίπεδο, ε, στο, επίπεδο, στο κατάλληλο επίπεδο σε σχέση με τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων. Και οι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικέ για τα θέματα αυτά. αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε τελική ανάλυση είναι σαφέ ότι ακόμα και αν έχουμε ξεπεράσει την κρίση Επιβίωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη χρηματοπιστωτικής κρίση παραμένουν πολλά τα οποία πρέπει να πράξουμε, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά ήδη και η σκληρή μα προσπάθεια αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Υπάρχει μια σημαντική μείωση στα spread μεταξύ των αποδόσεων των απολόγων των ομολόγων. Μια σύγκληση και μια ε, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ενίο νόμισμα είναι προαπαιτούμενο για την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και των καταναλωτών είναι απαραίτητο να προωθήσουμε και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, αλλά η σταθερότητα είναι προαπαιτούμενο για την ανάκαμψη. Πολλά έχουν επιτευχθεί μέσα στον τελευταίο χρόνο. Πριν από 12 μήνε ετέθη σε εφαρμογή το εξάπτυχο, το six pack. Και εφέτο δεχτήκαμε την, ε, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία για φιλόδοξε μεταρρυθμίσει στα κρατη που ήταν σημαντικό παράγον για την επιστροφή σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίση κατάφερε να τυθασεύσει την κρίση χάρη στις ενέργειές της και έχουμε φτάσει λοιπόν στα αποτελέσματα του τέλους του έτους για τα θέματα ε, τραπεζικής εποπτείας και για την βοήθεια προς την Ελλάδα. Το έχω πει και το ξαναλέω. Η πρόοδος μας είναι βήμα με βήμα πάντα. Αλλά αυτά τα βήματα συνεχίζουν. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει μια χρηματοπιστωτική κρίση τέτοιου μεγέθους. Τα εργαλεία αυτά θα έπρεπε να, έπρεπε να σχεδιαστούν, να τύχουν συμφωνίε, να εγκριθούν και πολλέ φορέ να κυρωθούν και από τα κράτη-μέλη. Εξακολουθεί να υπάρχει κάποια δυσφορία από ορισμένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει με κάποια βραδιπορία και κάποια κράτη-μέλη έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ για να πάρουν τι απαραίτητε δράσει μεταρρύθμιση των οικονομιών του. Συνεχίζουμε όμω και επιμένουμε στι προσπαθίε μα και πιστεύω ότι θα επιτύχουμε. Εγώ πιστεύω πάντα ότι η βαθμία πρόοδος είναι ο χρυσούς κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πρόοδος βαθμία αλλά όχι κλειδονισμή. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αντιμετώπισε και άλλα θέματα. Είχαμε συζήτηση κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ήδη από το 2008, όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα ήθελα να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ένας λόγος είναι το θέμα της ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, το οποίο έχει γίνει σοβαρότερο τα τελευταία χρόνια. Οι χώρες μας ε, αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες στη διατήρωση της ειρήνης στην γειτονία μας αλλά και πέραν αυτής τελευταίες επιχειρήσεις για αντιμετώπιση κρίσεων όπως στη Λιβύη απεκάλυψαν κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Και το οικονομικό πλαίσιο θα έλεγα μας πιέζει να αναπτύξουμε ικανότητες με πολύ αποτελεσματικό οικονομικά τρόπο. Πριν από τη συνάντηση κορυφής είχα ζητήσει τη συνάντηση του Δεκεμβρίου του 2013 να αφιερωθεί στα θέματα αυτά. Στόχος της συζήτησης αυτής είναι να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες και οι κατευθύνσεις για τις προσπάθειές μας. Σε πρακτικό επίπεδο ζητήσαμε επίσης από την κυρία Άστον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν προτάσεις. Επί τη βάση αυτών των προτάσεων και μετά από διαβουλεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν με τα κράτη-μέλη, θα παρουσιάσω τις προτάσεις στη συνάντηση του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2013. Είχαμε επίσης και ε, συζητήσεις για την κατάσταση στη Λιβύη, η οποία χειροτερεύει, μια κατάσταση η οποία μας προκαλεί ε, πολλές ανησυχίες. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί, έτσι ώστε να βοηθήσει την κατάσταση και να στηρίξει τους αμάχους. Υπάρχει ανάγκη έτσι ώστε να περάσουμε σε μια νέα πολιτική κατάσταση επίσης και για τη Συρία. Υποστηρίζουμε ένα δημοκρατικό μέλλον για τη Συρία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό σε όλες ε, τις μειονότητες. Εν πάση περιπτώσει, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια καλή θετική εβδομάδα στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζουμε πάντα σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ό,τι αναλαμβάνουμε σαν προσπάθεια έχει σαν βασικό στόχο να ξεπεράσουμε τα προβλήματα απασχόλησης και την ύφεση. Αλλά υπάρχουν περισσότεροι λόγοι να είμαστε πιο αισιόδοξοι από ό,τι τις τελευταίες εβδομάδες, αν και ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς και δύσκολος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπαρός, εξ της Κομισιόν, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Εξωτήμα μέλη, όταν σας απευθύνθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ε, αφαιρεθούμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήρε αποφάσει καθοριστικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καθορίσουν το μέλλον μα για τους ερχόμενε εβδομάδε, μήνε και χρόνια. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν ένα βήμα προόδου. Ο ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για τι τράπεζε, δίνει το σωστό σήμα για την ε, Τραπεζική Ένωση που σχεδιάζει το Συμβούλιο. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12 Σεπτεμβρίου για τον ενιαίο αυτό εποπτικό μηχανισμό οδήγησε στην ομόφωνη θέση του Συμβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου, μόνον τρεις μήνες μετά. Το Κοινοβούλιο, χάρη στους εισηγητές του, την κυρία Τάισεν και τον κύριο Γκίγκολτ, ε, εργάστηκε με μεγάλη ταχύτητα και επιμέλεια, ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει αμέσω. Αυτό δείχνει ότι σεβόμενοι πλήρω ε, την ε, μοναδική θεσμική μα διοργάνωση μπορούμε ω Ένωση να ακολουθήσουμε τι σωστέ πολιτικέ κατευθύνσει, τη σωστή στιγμή εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Ο ενιαίος επιτυχικό μηχανισμό είναι αναγκαία θεμελία για την ε, Τραπεζική Ένωση. Είναι το απαραίτητο συστατικό στοιχείο τη νομισματική Ένωση. Όμω, θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους και να συμφωνήσουν σε αυτό και τα 27 κράτη-μέλη εντός του πλαισίου της συνθήκης έτσι, θα φανεί ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της ενίσχυσης της νομισματικής ένωσης ε, και διατηρώντας την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Επίσης, επιτρέπει να υπάρξει άμεσα ανακεφαλοποίηση ε, των τραπεζών από τον μηχανισμό σταθερότητα. Έτσι θα πάψει ο φαύλο κύκλο μεταξύ των ε, τραπεζών και των κρατικών χρεών. Ήδη τον Ιούνιο του 2012 υπήρξε δήλωση από τη Σύνοδο Κορυφή και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσφατα έδειξαν ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για το θέμα αυτό, όσο δυνατόν συντομότερα, το πρώτο εξάμεινο του 2013, ώστε να υπάρξει νέο εποπτικό μηχανισμό άμεσα και να αρχίσει να λειτουργεί. Ενώ ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα θα μπορεί να ανακεφαλοποιήσει απευθεία τι τράπεζε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ολοκληρωθούν σύντομα οι διαπραγματεύσει επιτυχημένα για του κοινού τραπεζικού κανόνε και σε εθνικό επίπεδο και για τα επίπεδα εγγύηση των καταθέσεων. Οι προτάσει αυτέ βρίσκονται στον πυρήνα του ενιαίου εγχειριδίου για τους ε, τράπεζε και για του ε, κανόνε κανόνες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για του κανόνε που θα εφαρμόζουν οι εθνικοί υπόπτες. Ελπίζω να υπάρξει λοιπόν συμφωνία στι προτάσει αυτέ ω το δυνατόν συντομότερα. Ανακοίνωσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει νέα μέτρα για έναν ενιαίο μηχανισμό για τι τράπεζε και συμφωνήσαμε τα μέτρα αυτά να εξεταστούν από του συνομοθέτε τα σειρά προτεραιότητε και με σκοπό να εγκριθούν τα μέτρα αυτά εντό αυτή τη κοινοβουλευτική θητεία. Είναι ένα λογικό επόμενο βήμα αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να δημιουργηθεί βιωσιμότερο και δικαιότερο τραπεζικό σύστημα με έναν ενιαίο μηχανισμό επίλυσης των προβλημάτων, αντιμετώπισης της κρίσης, όπου θα είναι ανθεκτικό το τραπεζικό σύστημα και οι δυσχέρειες των τραπεζών θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα. Η Τραπεζική Ένωση είναι σημαντική ως ένα σύνολο, ενιαίο σύνολο μιας βαθύτερης και ισχυρότερης νομισματικής ένωσης. Ήδη έγιναν συζητήσεις για το απότερο μέλλον της Νομισματικής Ένωσης ε, με την έκθεση του ε, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες ώστε να υπάρξει ένα πρόγραμμα και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τι νέε προκλήσει η, Νομισματική Ένωση. Έτσι θέλουμε να καταρτήσουμε μια σειρά προτεραιοτήτων ε, σε επίπεδο δημοσιονομικού συντονισμού, νομισματικής ένωσης, ώστε οι εθνικές πολιτικές να βρεθούν στην καρδιά της εθνικής κυριαρχίας και να παραμείνουν εκεί. Ήδη την περασμένη εβδομάδα είπα ότι δεν περιμένω να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για το απότερο μέλλον τη νομισματικής Ένωση. Όμω οι συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδειξαν το πόσο πολύπλοκα είναι τα ζητήματα που συζητώνται. Και πραγματικά ο επίγον χαρακτήρα δεν γίνεται αντιληπτό με τον ίδιο τρόπο σε όλε τι πρωτεύουσε. Πρέπει όμω να αναζητήσουμε τη συνένεση για να προχωρήσουμε. Πέραν αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το ΤΟΥΠΑΚ, ε, τη δέσμη αυτή μέτρων, ω άμεση προτεραιότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποβάλει προτάσει για τον επόμενο συντονισμό εξάντε των μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα εργαλείο σύγκληση και συντονισμού ως ένα θέμα μείζονο ε, ενδιαφέροντο για όλε τι κυβερνήσει, όπω είχε ε, συζητηθεί και τι τελευταίε εβδομάδε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου ο πρόεδρο και εγώ ε, θα κληθήκαμε να κάνουμε προτάσει για μέτρα για το τραπεζικό σύστημα και για το εφικτό των ε, συστημάτων, των συμβάσεων αυτών που θα επιτρέψουν ε, στην, ε, στις τράπεζες να ενισχυθούν. Τέτοια εργαλεία και τέτοιοι μηχανισμοί πρέπει να ταιριάζουν και με το πλαίσιο των ευρωπαϊκών συνθήκων, του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονήματο και τη δημοσιονομική διοργάνωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τι υπάρχουσε διαδικασίε πρέπει να κινηθούμε και για το μέλλον, χωρί να αναζητούμε επιπλέον επίπεδα διακυβέρνηση. Να εντοπίσουμε εξειδικευμένε προκλήσει που πρέπει να, αντιμετωπιστούν. Κάτι δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένε πιέσει. Ένα τέτοιο εργαλείο που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη ε, να αντιμετωπίσουν ειδικέ ανάγκε και ειδικέ ελλείψει ισορροπία. Πρέπει να δούμε εδώ και το θέμα τη ανταγωνιστικότητα, που θα ήταν μια περαιτέρω συμβολή στον κατάλογο προτεραιοτήτων μα για την ανάπτυξη γιατί θα πρέπει εδώ να συνδυάσουμε οπωσδήποτε και αυτό το σκέλο, την ανάπτυξη με την ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε μια συνολική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κοινοτική μέθοδο και βεβαίω υπό τον έλεγχο και την κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόθεσή μα είναι να υποβάλουμε νέε ιδέε μετά την απόφαση για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά τι διαβουλεύσει βεβαίω που θα έχουμε μεταξύ των θεσμικών οργάνων και με το δικό σα σώμα θα πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στην Ένωση ώστε να λάβουμε ευρείε πολιτικέ αποφάσει, συμπεριλαμβάνοντα τα περισσότερα ζητήματα που μα απασχολούν, όπω το αποτύπωμα τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν θα αποκλεί βεβαίω ε, μελλοντικέ αλλαγέ στο μέλλον εφόσον χρειαστούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν ε, συμφωνήσει σε ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο. Όμω έχουμε γοργέ εξελίξει και θα πρέπει, όπω προτείνεται και στο αποτύπωμα αυτό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχουμε και βαθύτερε συζητήσει και σε επίπεδο κρατών μελών. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την κοινωνική διάσταση, τη σημασία τη κοινωνική διάσταση τη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, συμπεριλαμβάνοντα εδώ και τον κοινωνικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται στην θεσμική διοργάνωση τη Νομισματική Ένωση και όλοι έδωσαν έμφαση στο να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία σε όλε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, με κοινέ δράσει σε εθνικό επίπεδο, ώστε να θεμελιώδη ζητήματα ισότητα και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη να διασφαλίσουμε την δημοκρατική νομιμότητα και τη λογοδοσία, ενώ επιτελούμε πρόοδο στην Νομισματική Ένωση, είναι προτεραιότητα και αυτό φάνηκε και στην ε, πρόσφατη έκθεση τη Προεδρία και στο αποτύπωμα τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, δήλωσε ότι η περαιτέρω σύγκληση της, του σχεδιασμού πολιτική και ο συνδυασμό των πόρων πρέπει να συνοδευτούν από την πλήρη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου. Αγαπητά μέλη, την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε για τα θέματα αυτά και στα πλαίσια της ετήσιας ε, μελέτης για την ανάπτυξη και συμφώνησε σε πέντε προτεραιότητες που πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εξετάσει το, τη δέσμη μέτρων του AGS ε, μέχρι την Εαρινή Σύνοδο και τα συμπεράσματα καλείται το Συμβούλιο να ε, υποβάλει δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων με σκοπό να υιοθετηθούν οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συστέσει και για εγγυήσει προ την όλια ε, με απότερο ορίζοντα το 2014. Αυτό το καλωσορίζουμε. Εάν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη που να προσφέρει θέσει εργασία και να αντιμετωπίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα πρέπει να διασφαλίσουμε στου νέου την εκπαίδευση, την ε, κατάρτιση και ότι βεβαίω θα μπορούν να ζητήσουν καλύτερη εργασία και με μεγαλύτερο χρονικό ρίζοντα από τέσσερι μήνε. Η ανάκαμψη βεβαίω απαιτεί να αξιοποιήσουμε όλε μα τι δυνατότητε, την ενιαία αγορά δηλαδή. Οι συνομοθέτε θα πρέπει να ολοκληρώσουν τι συζητήσει για τα μέτρα που προκύπτουν από την πράξη για την ενιαία αγορά, την πρώτη πράξη για την ενιαία αγορά. Εδώ πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσουμε ότι τα 7 μέτρα προτεραιότητα θα εγκριθούν και θα υλοποιηθούν ω τα δυνατόν συντομότερα. Σε ό,τι αφορά την ε, δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά, θα πρέπει μέχρι το Μάρτιο του 2013 να έχουν υποβληθεί νέε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υιοθετηθούν στον επόμενο κύκλο εργασιών του Κοινοβουλίου. Εδώ θα είναι ψηλά ο πύχη των προσδοκιών και των απαιτήσεών μα, ε, απαιτώντα αλλαγές και σε ευαίσθητους τομείς, όπως στις τεχνολογίες δικτύου και δικτύωσης. Νομίζω όμως ότι και σε κυβερνητικό επίπεδο υπάρχει μια νέα δέσμευση προς την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ευφυή νομοθεσία. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να επιταχύνουμε την πρόοδο. Και βασιζόμενοι σε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε εν τέλει να συμφωνήσουμε στο ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρυστεχνία. Μετά από 30 χρόνια ήρθε επιτέλου η στιγμή να γίνει και αυτό. Αγαπητά μέλη, στο Συμβούλιο έγιναν και σημαντικές συζητήσεις για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα θέματα άμυνας. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κ. Βαν Ρόμπαϊ. Να πω όμως ότι η συνάντηση κορυφής αυτή ήταν μια συνάντηση με πολλή δουλειά, ίσως όχι με μεγάλους πρώτους τίτλους εφημερίδες. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν αυτές οι μεταρρυθμίσεις να τις νιώσουμε ότι ανήκουν σε όλες μας σε εθνικό επίπεδο. Έτσι θα εμβαθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να δείχνει την φιλοδοξία η οποία είναι απαραίτητη. Αυτή η φιλοδοξία θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω αποφάσεις πέραν αυτών οι οποίες ήδη ελήφθησαν όπως για το SSM και μετά υπήρξε και η συμφωνία για την Ελλάδα. Αυτά δείχνουν ότι ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε την κρίση και ταυτόχρονα έχουμε και μακροπρόθεσμες προοπτικές και οράματα. Μπορούμε να ξεπεράσουμε τις παρούσες δυσκολίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα, να προχωρήσει με τις προτάσεις που ήδη ανακοίνωσε και ελπίζω να συνεχίσουμε τις προσπάθειες το 2013. Πρώτη προτεραιότητα θα είναι το ταχύτερο δυνατόν να καταλήξουμε στο MFF δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο προπολογισμό μα, ο προπολογισμό τη Ένωση, είναι ένα προπολογισμό ανάπτυξη και ένα δημοσιονομικό πλαίσιο πολιετές είναι απαραίτητο για να υπάρξει ανάπτυξη. Θα κλείσω εδώ ευχαριστώντας σας όλους, ελπίζω να έχετε καλές γιορτές, να ξεκουραστείτε και η επόμενη χρονιά να είναι μια πολύ εργατική χρονιά. Ο κύριος Γιώσεφ Τόλα από την ομάδα του ΕΛΚ έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας έχει εγκρίνει τον ενιαίο μηχανισμό τραπεζικής εποπτείας SSM και έχει δημιουργήσει και τις βάσεις για μια τραπεζική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός και είμαι ικανοποιημένος γι' αυτό, αλλά φυσικά δεν, δεν επαρκεί. Η πολιτική των βημάτων προς τα εμπρός έχει νόημα μόνο όταν βρίσκεται μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Και επίσης όλα αυτά τα οποία αποφασίζονται πρέπει να εφαρμόζονται και να προχωρούμε περισσότερο. Αλλιώς θα βρούμε ότι υπάρχουν τρύπε στο δίκτυ. Υπάρχουν τρύπε οι οποίες θα αφήσουν ορισμένες τράπεζες να εκφύγουν από το σύστημα εποπτείας. Να μην ξεχάσουμε τα διδάγματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όλες οι τράπεζες πρέπει να τη χάνουν απαραίτητες και δε, φυσιολογικά δεν πρέπει να έχουν να αποκρύψουν τίποτα. Λέτε ότι μια τράπεζα αρκεί να αποτύχει για να κλειδονιστεί το νέο σύστημα το χρηματοπιστωτικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την ταχεία υιοθέτηση ενός κοινού κανονισμού ο οποίος θα εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες όλων των κρατών μελών. Και είμαστε πεπισμένοι επίσης ότι πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στην ενίσχυση οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το εξάπτυχο, το ΣΕΚΣΠΑΚ, να δώσουμε έμφαση στη σταθερότητα, τον συντονισμό και την διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει κάτι επιγόντως να έχουμε μια συμφωνία για το δίπτυχο, το ΤΟΥΠΑΚ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να πω ότι αρχίζω να κουράζομαι να ακούω τα ίδια πράγματα. Και βλέπω και σε εσά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φανεροπάκη, κύριε Μπαρόσο, μια κάποια κόπωση. Το μήνυμά μου είναι πάντα το ίδιο. Γνωρίζουμε ποιε είναι οι λύσει οι οποίε πρέπει να υλοποιηθούν και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ληφθούν οι αντίστοιχε αποφάσει. Θα πρέπει να έχουμε όμω το θάρρο να πράξουμε τα απαραίτητα. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μονάχα τι επικείμενε εκλογέ, να είμαστε όμως πολιτικοί που σκέφτονται για το μέλλον και τις επερχόμενες γενναίες. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την πολιτική ως σοου. Ορισμένοι ήδη θέλουν να επιτεθούν κατά της Ευρωπαϊκής Δημοσίας Διοίκησης. Εγώ δεν δέχομαι αυτήν την αντιμετώπιση. Έχουμε υπηρεσίες ποιότητας που εργάζονται κάθε μέρα για την Ευρώπη και για το μέλλον της Ευρώπης. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους πριν από τα Χριστούγεννα και αυτοί οι οποίοι θέλουν να συκοφαντήσουν αυτήν την δημόσια διοίκηση, θέλουν να καταλύσουν την ευρωπαϊκή ενωσιακή αντιμετώπιση για να προκρίνουν την διακυβερνητική διαδικασία. Γιατί οι υπάλληλοι των κρατών μελών πληρώνονται εξίσου καλά με τους ευρωυπαλλήλους. Και τα γνωρίζετε αυτά πολύ καλά. Ξέρετε ποια είναι η σύγκριση μεταξύ των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διακυβερνητικών υπαλλήλων. Εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φυσικά πρέπει να υπάρχει και κάποια εποπτεία για όλα αυτά τα θέματα. Πολλέ φορέ είναι οι ίδιοι οι οποίοι επιτίθενται στου ευρωπαϊκού θεσμού και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν ένα αποτελεσματικό προπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πολιτέ πλαίσιο για τα δημοσιονομικά το οποίο προτείνει η Κομισιόν είναι περισσότερο από απαραίτητο. Θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει των 7 επερχομένων ετών και το σχέδιο εργασία είναι η κατεύθυνση προ την οποία πρέπει να κινηθούμε. Όπω είπατε, κύριε Φανρομπάη, χρειαζόμαστε κατευθυντήρε γραμμέ, σαφέ χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Με του απαραίτητου κανονισμού και οδηγίε έγινε δυνατό να έχουμε μια ενιαία αγορά το 1992. Σήμερα είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση και συγχρόνω να ενισχύσουμε την νομιμοποίηση και την υπευθυνοποίηση που πρέπει να συνοδεύουν αυτή την ενιαία αγορά. Και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι ο καλύτερο εγγυητή για κάτι τέτοιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι εθνικέ λύσει είναι καλύτερε και πιο σημαντικέ από την ενωσιακή, σα ρωτώ, τι φοβόσαστε. Η Ευρώπη έχει εξασφαλίσει την ειρήνη και την ευμάρεια και την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είτε πρόκειται για τον αγώνα κατά των ανισοτήτων, την ενίσχυση των υποδομών, την τροφιμική ασφάλεια, την ποιότητα του περιβάλλοντος, την παιδεία και την κατάρτιση, η Ευρώπη είναι υπόδειγμα και φάρος για τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα όμως χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε και πάλι την πεποίθησή μας σε μια πολιτική Ευρώπη. Αυτή είναι μια ευχή που κάνω για το νέο έτος, που πρέπει να ξεπεράσει τους επαναληπτικούς λόγους και πρέπει να μας οδηγήσει να εστιάσουμε στα ουσιαστικά μια πραγματική νομισματική, οικονομική και πολιτική ένωση. Ξέρω ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν συμμερίζονται μια τέτοια κατεύθυνση και μιλάνε ακόμα και για να, για να το ξαναδιαπραγματευτούν την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σέβομαι τη θέση αυτή και για να είμαι ειλικρινής, εγώ λυπήθηκα όταν άκουσα ότι ο Ντέβιτ Κάμερον αποφάσισε να μην είναι παρόν στην απονομή του βραβείου Νόμπελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έτσι ο Βρετανικός, ο Βρετανός ε, Πρωθυπουργός δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το ρόλο της Αγγλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Winston Churchill και τον περίφημο λόγο του. Έχουμε το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φέρει το όνομά του. Ο Winston Churchill υποστήριξε και αυτό στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και την ε, κοινή δράση. Και ο Edward Heath, η Margaret Thatcher που, υπογράμμισε την, που υπέγραψε την κοινή πράξη και ο John Major που υπέγραψε τη συνθήκη του, του Για όλους αυτούς τους Άγγλους πολιτικούς έχω μια τεράστια, ένα τεράστιο θαυμασμό και ε, εκτιμώ το έργο τους. Δεν είμαι αντιβρετανικός, αλλά ως πεπισμένος ε, Ευρωπαίος δεν μπορώ να δεχτώ τη λογική της Βρετανικής κυβέρνησης, γιατί έχει περάσει από την προηγούμενη στάση της σε μια στάση η οποία δεν μου φαίνεται πραγματιστική. Γιατί ψηφίζει κατά του ετήσιου προϋπολογισμού του ετήσιου προϋπολογισμού γιατί θέλει επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουν οι Βρετανοί να ξαναδιαπραγματευτούν, γιατί αυτό πρέπει να μα εμποδίσει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει πάντα τα κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι να μπορούν να αναδιαπραγματευτούν τη θέση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να τροχοπεδεί τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και επίση θα ήθελα να κατανοήσω το lobbying που γίνεται, την πίεση που γίνεται για να υπάρχουν θέσει γενικών γραμματέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιδίω στου τομεί που επιμένει το ευρωπαϊκό το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εκεί πρέπει να διευκρινιστεί η κατάσταση. Εγώ δεν θέλω να είμαι επιθετικό. Θέλω απλώ να διευκρινιστούν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα κοινή λογική. Πρέπει να τεθούν όλα επιτάπητο και να συζητηθούν από κοινού μαζί με τη συζήτηση του ε, προπολογισμού του 2013 και του πολιετού πλαισίου. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει. Ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να προχωρήσουμε ω 27 κράτη και 28 αύριο μαζί με την Κροατία Ας σκεφτούμε λοιπόν τους μεγάλους ηγέτες της Ευρώπης που είχαν το θάρρος να προωθήσουν την Ευρώπη γιατί ξέροντας ότι η περισσότερη Ευρώπη είναι προσθέμενη αξία και για τις δικές τους χώρες και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και με την ευκαιρία αυτή σας εύχομαι χαρούμενα και ειρηνικά Χριστούγεννα και νέο έτος και ελπίζω ότι με το νέο έτος θα επανέλθετε με ενεργητικότητα στην προσπάθεια να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. <clears throat> Για τους ε, Ισπανούς για Σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Σαλόμ Γκερέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας μας είπατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια καλή εβδομάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ εν μέρει μαζί σας. Αλλά νομίζω ότι ήδη το ότι υπήρξε και μια καλή εβδομάδα είναι ένα μεγάλο νέο και αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος Μπαρόσο είπε επίσης ότι ε, και θα συμφωνήσω μαζί του ότι δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Ε, κάτι βέβαια το οποίο δεν σημαίνει ότι στο παρελθόν τα πράγματα ήταν πάντα καλύτερα. Υπάρχουν θετικές πλευρές, αλλά θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τους κινδύνους, τις ανεπάρκειες, τις δυσλειτουργίες οι οποίες παρεμποδίζουν τη σωστή εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς θεωρώ ότι η έγκριση του ενιαίου μηχανισμού υποπτία είναι ένα θετικό βήμα είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα. Είναι ένα βήμα το οποίο ανταποκρίνεται με τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει το Κοινοβούλιο μας με πάρα πολύ ψηλή ταχύτητα και με πολύ μεγάλη προσπάθεια μέσω των δύο εκθέσεων τις οποίες έχει εγκρίνει, Tyson και Giggold. Ο μηχανισμός θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις δυνατότητες εποπτείας. Θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στα πιστοτικά ενδρύματα ε, και σωστή ενημέρωση μέσω των, εθνικών, των ε, κεντρικών εθνικών τραπεζών. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο κείμενο, όπως είπε ο κύριος Μπαρόσο, έχουν, ε, θα συνεχιστούν οι, πραγμα, οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για τα θέματα αυτά. Πάντως υπάρχει όχι ιδιαίτερα πολύ μεγάλη ευκρίνεια στο πώς θα τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός της τραπεζικής εποπτείας και το εάν αυτή η θέση σε λειτουργία θα δώσει πραγματικά τη δυνατότητα να υπάρξει θα έλεγα ανακούφιση ε, στα χρέη των τραπεζών και ανακούφιση του δημοσίου χρέους σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να είναι λειτουργικό το σύστημα και απαιτείται χρόνος για να επιληθούν ορισμένα προβλήματα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτό που είναι σαφές είναι ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήμασταν ιδιαίτερος φιλόδοξοι και πιστεύαμε ότι το πλαίσιο δυνατότητας παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είναι σήμερα. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε και με τους άλλους δύο πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης. Νομίζω ότι για τα οικονομικά θα πρέπει τα οικονομικά ιδρύματα να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών και θα πρέπει επίσης η προσπάθεια αυτή να γίνεται από τον ίδιο τον πιστοτικό τομέα. Το σύστημα των εγγυήσεων των καταθέσεων λυπούμεθα αλλά σε αυτή τη φάση έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Υπάρχουν όμως και ορισμένες ανησυχίες. Έχουμε καταρχάς... Ε, Μια μεγαλύτερη σύγχυση σε λειτουργικό επίπεδο. Μας παιδί η καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Εξακολουθεί να υπάρχει η προσέγγιση μόνο της εδραίωσης των δημοσιονομικών και όχι η ανάπτυξη και η απασχόληση, όχι η αηφορία σε κοινωνικό επίπεδο. Και υπάρχει και μια αντίδραση και αντίσταση στο δημοκρατικό έλεγχο που πρέπει να ασκείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει αυτή η σύγχυση. Ο ίδιος ο κύριος Σούλς στην αρχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι ήδη είναι πάρα πολύ πολύπλοκη η θεσμική μας αρχιτεκτονική και αρχίζει πια να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το δίπτυχο, το εξάπτυχο, τις συμφωνίες μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών, τα συμβόλαια ανταγωνιστικότητας, όλο και περισσότερο με το Jacques Delors που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα, ε, μη, μη αναγνωριστό πολιτικό αντικείμενο, ένα είδος πολιτικού ούφο. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την σαφήνεια για τους πολίτες μας που είναι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η βραδιπορία. Πολλά από αυτά τα οποία γίνονται σε κάθε συμβούλιο αναβάλλονται για το επόμενο Συμβούλιο του Ιουνίου του 2013, μετά από έξι μήνες. Όπως είπε ο κ. Βαν η βαθμία προσέγγιση και όχι οι απότομες αποφάσεις είναι τμήμα της παράδοσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν διαφορετικές μορφές βαθμίας προσέγγισης. Οι κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις κάθε εβδομάδα σχεδόν, εμείς κάθε έξι μήνες. Εμείς έχουμε ένα ορίζοντα ενός, ενάμιση έτους μέχρι το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα που μας ξεχωρίζει από τα κράτη-μέλη. Και είναι άτολμη η προσέγγιση μας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στη δεύτερη μου παρέμβαση θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Υπάρχει μια ουσιαστική αδυναμία σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα, τον κοινωνικό πυλώνα, που είναι η βάση, το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε μονάχα μια οικονομική και νομισματική ένωση, είμαστε ένα πολιτικό εγχείρημα που πρέπει να έχει μια βάση στην αγορά, στην νομισματική ένωση, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να βασίστε σε ένα σύνολο αξιών, σε ένα κοινωνικό μοντέλο, στην κοινωνική, στην ε, δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Και αυτή η δημοκρατική συμμετοχή θα πρέπει να εκφράζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αποφάση λοιπόν του Συμβουλίου σε σχέση με την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση είναι ένα άτολμο βήμα, ένα βήμα το οποίο δεν θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τη σωστή σύνδεση και συνεργασία των θεσμικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεργασία που είναι απαραίτητη για να γίνει σεβαστή η κυριαρχία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Κοινοβουλίου μας. Ευχαριστώ, λέει ο Σας ευχαριστώ κύριε Βιγερέρο. Για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Φερχόφστατ. I think that we have to be honest, European Council. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια φορά το έσωσαν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομία και Οικονομικών. Διότι χωρί τη δική του συμφωνία και τη συνένεση δεν θα, υπήρξαν τόσο, δεν θα υπήρχαν τόσο πολλά να, ε, για τα οποία να πανηγυρίζουμε σήμερα. Είπε ο κύριο Μπαρόζο ότι όλε οι επιλογέ είναι ανοιχτέ. Δηλαδή δεν υπάρχουν συμπεράσματα στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένα χειροπιαστά συμπεράσματα. Ξανάρθουμε όμω τη θετική διάσταση αυτού του Συμβουλίου. Την ε, συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων Υπουργών ε, Οικονομικών. Νομίζω ότι ο νέο εποπτικό μηχανισμό για τις τράπεζες είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο, ο εποπτικός αυτός Έλεγχο μηχανισμό ήταν από τι αρχέ του 2009 και 2010 η θέση του Ευρωκοινοβουλίου. Το θυμάστε το πακέτο για την εποπτεία. Το λέγαμε για μήνε και μήνε. Ενιαίο επόπτη θέλαμε. Και ε, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου μα λέγανε όχι, όχι. Δεν είναι η στιγμή να γίνει αυτό. Με την ενδιάμεση αναθεώρηση. Να λοιπόν που πριν από αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση έχουμε τον ενιαίο επόπτη. Διότι προφανώ ήταν σωστή η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Καλά κάναμε και επιμέναμε πριν από δύο χρόνια γι' αυτό. Όμως δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Μόλις τώρα αρχίζουν οι πραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το θέμα. Μισό, ε, το μισό από τη δέσμη, μισή από τη δέσμη αυτή μέτρων θα πρέπει να περάσει τη διαδικασία της ε, σύνομοθεσίας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά τη συμφωνία των ε, Υπουργών Οικονομικών για συγκεκριμένα σημεία ένα ενίο επόπτη θα εποπτεύει μέρη, τμήματα τη ενιαία αγορά ή συνολικά την ενιαία αγορά. Επίση, τι κίνητρα θα έχουν οι χώρε εκτό του συστήματο, τουλάχιστον στην αρχή, να συμμετάσχουν σε αυτό το σύστημα τη ενιαία εποπτεία. Μήπω στο μέλλον δημιουργήσουμε μια κατάσταση, μια δικασία διπλή διδιοταχυτήτων ως προς την ε, ε, εποπτεία. Μήπως δημιουργούμε ένα συνικό τείχος, ένα ξεπέραστο εμπόδιο δηλαδή, την δημοσιονομική εποπτεία από τη μία και την τραπεζική εποπτεία από την άλλη. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ γραφειοκρατικό το σύστημα, γεμάτο παραθυράκια και θα έχει πάρα πολλή δουλειά το Κοινοβούλιο να κάνει για να διορθώσει τις προτάσεις που έχουμε τώρα στα χέρια μας. Ώστε εν τέλει να μην λειτουργεί σε επίπεδο μελών το σύστημα, αλλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό δεν είναι τώρα καθόλου σαφέ στην τελική συμφωνία των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τα λοιπά στοιχεία τη συμφωνία. Λυπάμαι, αλλά δεν έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ. Ε, με συγχωρείτε που είμαι τόσο ε, Όμω, αλλά δεν μπορώ να συμμεριστώ τη δική σα ε, την χαρά κύριε Φανρόμποη. Αν διαβάσετε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, το σημαντικότερο, το ζωτικότερο στοιχείο για τη νέα Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν αναφέρονται. Έχουν παραγωνιστεί τελείως στο αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται και στο έγγραφο του Κοινοβουλίου, αλλά όχι στα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει τίποτε ούτε για το Ταμείο Διάσωσης, ούτε για την ε, εγγύηση για τα χρέη για την κοινή ανάληψη του χρέους. Δεν υπάρχει κανένα, ε, καμία αναφορά για το Κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο, για τις δημοσιονομικές δυνατότητες, τις ιδέες αυτές για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, τα βήματα προόδου που θέλαμε για να προχωρήσουμε με το ευρώ. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά κύριε Μπαρόζο, όπως είπατε. Εγώ τα βλέπω διαφορετικά βέβαια από εσά, όχι με αισιοδοξία, διότι αν δεν υπάρχουν αυτέ οι μνήμε στα συμπεράσματα που πήγανε. Εγώ τουλάχιστον έτσι ερμηνεύω το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν ασκείται πίεση προ του ε, πολιτικού αρχηγού ε, τη Ευρώπη να λάβουν αποφάσει για την νομισματική ε, και οικονομική ένωση. Και ο λόγο είναι σαφή. Οι εκλογέ στη Γερμανία το Σεπτέμβριο μπλοκάρουν τα πάντα. Εντάξει, το, περι... το καταλαβαίνουμε. 9 μήνε να περιμένουμε και δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο το διάστημα. Και για μια πολιτική σταδιοδρομία μικρό είναι ω χρόνο. Το ξέρετε κύριε Πρόεδρε. Σας βλέπω που σημειώνετε στο χαρτάκι σα. Είναι προσωπικέ σημειώσει, βέβαια, αλλά Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι ο πραγματικός λόγος που δεν φαίνεται να υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη είναι οι ε, αποφάσεις του κυρίου Ντράγκη. Ο κύριος Ντράγκη επελέγει χθε ως άνθρωπος της χρονιάς από τους Financial Times και έχει κάνει τεράστιο έργο, όντω. Ε, βραχυπρόθεσμα την αναχέτησε την κρίση, αλλά μακροπρόθεσμα δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι καλό δεν ασκείται πλέον πίεση στους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων να προχωρήσουν με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ο κύριος Ντράγκη βρίσκεται και αυτό σε αδιέξοδο. Ζητά περισσότερη φιλοδοξία από τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ταυτόχρονα η δική του η φιλοδοξία έχει περιοριστεί. Είναι θεμελιώδες φάλμα να πιστεύουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι η κρίση έχει ξεπεραστεί θα χρειαστεί να δούμε ξανά τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Φερχόφσταντ για τους πράσινους. Έχει το λόγο η κυρία Ρεμπέκα Χάμς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και το Συμβουλίο και την Κομισιόν για την παρουσίασή σας. Έχει καταστεί δηλαδή ήδη σαφές να εξασφαλίσουμε χωρίς μεγάλες αντιπαραθέσεις μια πραγματική λειτουργική αρχιτεκτονική για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι υπάρχει η απαρχή μιας διαδικασίας ευρωπαϊκοποίησης των μεγάλων τραπεζών, γι' αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Τα μεγάλα κράτη, ακόμα και η περήφανη Γαλλία, έχουν αποδεχθεί το γεγονός ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες βέβαια να ρυθμιστούν, αλλά κατά την άποψή μου η Τραπεζική Ένωση θα είναι το αποφασιστικό βήμα το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κύριος Φερχόφστατ έχει δίκιο σε πολλά πράγματα και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στους προέδρους, τον κύριο Μπαρόζο και στον κύριο Φαν και θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Φερχόφστατ με κίνδυνο να σας κουράσω. Θα πρέπει να σκεφτείτε καλύτερα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο που είναι η πιο ισχυρή και η οδηγούσα δύναμη που θα επιτύχει τη μεγαλύτερη εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτό το ρόλο. Θα πρέπει να θυμηθείτε ότι προώθησε την νομοθεσία για το εξάπτυχο και το δίπτυχο και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι αυτό το οποίο θα διαδραματίσει τον κεφαλαιόδη ρόλο για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο το ζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και το οποίο οι αρχηγοί κρατών μελών και κυβερνήσεων το έχουν σπρώξει πέραν του, Ορίζοντο του ορίζοντος και αυτό δεν αναφέρομαι μόναχα για τη Γερμανία. αναφέρουμε σε πολλές άλλες χώρες που έχουν πάρα πολλές ανησυχίες και αμφιβολίες και αυτό φάνηκε και από την ηλιοτυπία που παρουσίασε ο κ. Φάνου Ρομπάι για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια νέα α, συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, όχι ξαφνικά αλλά μετά από πολύ καλή προετοιμασία. Είναι πραγματικά δικός μας, δικό μας καθήκον να μην σκεφτόμαστε για την Ευρώπη μόνο όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπαρόσο, αλλά ήδη προηγουμένω εμεί θέλουμε να εξηγήσουμε στου πολίτε γιατί θέλουμε εμεί περισσότερη Ευρώπη, γιατί θέλουμε να τεθεί από κοινού το χρέο των κρατών μελών, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μια αμοιβαία υπευθυνότητα και μία αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας υπουργό Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό <clears throat> για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες θα είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτή την τρομερή ανεργία που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει μονάχα να αντιμετωπίζει με ευχές το Συμβούλιο και την Κομισιόν να του απευθύνει ευχές, αλλά θα πρέπει να έχει την ευκαιρία μέσα από μια συνέλευση να συμβάλλει στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν είναι κατανοητή αυτή η θέση, τότε θα πρέπει να γίνει εν καιρό και αυτή η συνέλευση. Ευχαριστώ για, του... για τους συντηρητικούς. Έχει το λόγο ο κύριος Έπινγκ. Κύριε Πρόεδρε, τα αποτελέσματα του πλέον πρόσφατου Συμβουλίου μου θυμίζει τον ποιητή Αλεξάντερ Πόπου, ο οποίος ε, είχε γράψει σε ένα δοκίμιο του ότι εκεί όπου δεν τολμούν να πάνε οι άγγελοι, ορμούν οι παρανοϊκοί. Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα εδώ να ακούσω με συμπάθεια αυτά που είπατε, αλλά ε, θα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Ως εκ τούτου λοιπόν η συνάντηση αυτή στην οποία παρίσταστε ήσαν, ήταν μια συνάντηση αγγέλων από ό,τι φαίνεται. Έχετε προχωρήσει σε μέτρα για τις πιστοτικές δραστηριότητες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε αρμοδιότητες, υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα, ακόμα και ο αριθμός των τραπεζών που θα πρέπει να υποπτευθούν έχει καθοριστεί. Τέθηκαν τα θεμέλια λοιπόν δεύτερον θα υπάρξει ένα ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτεί ο ίδιος ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Καλό είναι αυτό, συμφωνώ με αυτό, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα χρήματα των απλών πολιτών. Τώρα όμως από εδώ και πέρα έρχονται και οι παρανοϊκοί στην περίπτωση. Καταρχάς το σύστημα εγγυήσεων, η αποταμίευση των πολιτών σε μία χώρα θα πρέπει να χρηματοποιούνται σε χώρες οι οποίες έχουν σορεύσει ε, χρέος σε άλλες χώρες. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη, είναι απρόσεκτη συμπεριφορά των τραπεζών. Και επίσης κάποιοι θέλουν να δημιουργηθούν και τα λεγόμενα ομόλογα τύπου γκουλάγκ λέει ο μιλητής. Κακή ιδέα. Γιατί κάποιοι οι οποίοι ε, πληρώνουν ακριβά τον δανεισμό τους, ε, πληρώνουν φυσικά περισσότερο από άλλους που πληρώνουν ευθυνότερα. Αυτό δεν είναι θέμα αλληλεγγύης, είναι κάτι το οποίο σαν διαφορά έχει αρχίσει από ό,τι φαίνεται να αντιμετωπίζεται. Ε, κάποιοι λένε ότι ε, θα είναι αντίθετοι με τη δημιουργία των ε, ευρωπαϊκών ομολόγων όσο ζουν. Τους εύχομαι φυσικά μια ιδιαίτερος μακρά επιβίωση στην ζωή αυτή. E Ευχαριστώ για την ομάδα Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Χέλμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε το μηχανισμό σταθερότητας, είχαμε δανειοδότηση, είχαμε διασφαλίσεις και τώρα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και οι σύμβουλοι της Deutsche Bank λένε ότι δεν υπάρχουν γερά θεμέλια για αυτά. Όπω και αν έχει, καμία από αυτές τις πρωτοβουλίε δεν έχει αντιμετωπίσει τις βασικές ελλείψεις ισορροπίας που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Πώς μπορεί κανείς να φανταστεί ότι η κοινή τραπεζική εποπτεία θα αντιμετωπίσει την ελληνική ανταγωνιστικότητα ή τα πλεονάσματα, τα, τα πλεονάσματα του εμπορικού ισοζυγίου στη Γερμανία. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να λυθεί το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, οι βασικέ, οι σταθερέ και μαζικέ ε, δημοσιο δημοσιονομικές μεταφορές. Ήδη από το 1997 είχαμε πει ότι για τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη χρειάζονται τέτοιες μόνιμες μεταφορές 6-8% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτή αγνοήθηκε ως προτροπή και βλέπετε τώρα τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως τέτοιες ε, μεταφορές ποσών θα ήταν προφανώς απαράδεκτες για τους Γερμανούς ψηφοφόρους. Έπειτα θα μπορούσαμε να δεχτούμε την επιλογή της ε, πτώχευσης. Να υπάρξει υποτίμηση δηλαδή και αποπληθωρισμό στην Νότια Ευρώπη. Όμως τέτοιο δεν μπορεί να το αντέξει το δημοκρατικό μας πλαίσιο. Οι Έλληνες ψηφοφόροι δεν θα μπορούσαν να το δεχτούν ή θα μπορούσε να, συμβεί, να, γίνει προφανής επιλογή. Να διαλυθεί η Ευρωζώνη, να επιτραπεί στην Ευρώπη να πτωχεύσει, να υποτιμήσει το νομισμά της, να ξαναγίνει ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές, να αρχίσει να μπορεί να είναι εμπορική για τις ε, θέσεις απασχόλησης και την ευημερία. Όμως το πολιτικό <coughs> κεφάλαιο που έχετε επενδύσει σε αυτές τις πρωτοβουλίες σας είναι τεράστιο. Δεν μπορείτε να παραδεχτείτε ότι κάνετε λάθος. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Φαρόμποε, κύριε Σούλτς, δική σας είναι η ανοησία. Δική σας είναι η έλλειψη ευθεία για την εξέβρεση λύσης. Εδώ όμως φαίνεται ότι ενώ η Αθήνα πεινάει, εσείς ε, τραγουδάτε το δικό σας, ε, το δικό σας χορό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ καλά τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουμε τέτοιους ε, δισταγμούς. Δεν βλέπω γιατί ο κύριος Ντόλ δυσκολεύεται να καταλάβει τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ντόλ, με μεγάλη χαρά να σας εξηγήσω τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ για την ομάδα της ενιαίας αριστεράς, ο κύριος Λεγιάρικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για, την, ε, για τα πεπραγμένα που μας αναφέρατε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φοβάμαι όμως ότι δεν υπάρχει συνολικό όραμα, δεν υπάρχει ένα σχέδιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα μας επέτρεπε να εξέλθουμε από την κρίση τη στιγμή που υπάρχουν τόσα σχέδια για απολύσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οποία δεν είπατε τίποτα, τη στιγμή που υπάρχει αύξηση τη ένδυα και πάλι δεν είπατε τίποτα, τη στιγμή που είναι υποχρεωμένα όλα τα κράτη να μειώσουν τους προϋπολογισμούς τους. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται μια φυγή προς τα πρόσω σε αυτή την κρίση. Γιατί δεν υπάρχει μια συνέχεια αυτών που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου που είχε αποφασίσει για ένα προϋπολογισμό 120 δισεκατομμύριων ευρώ. Αλλά δεν μας είχε πει τι θα χρηματοδοτηθεί, πόσες θέσεις εργασίας ή καταργήσεις θέσεις εργασίας μπορούν να αποφευχθούν. Σήμερα το νέο σχέδιο είναι ο μηχανισμός τραπεζικής εποπτείας. Προφανώς είναι απαραίτητη αυτή η εποπτεία. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι και διάδικος και δικαστής. Εάν πρόκειται για το θέμα της εποπτείας, γιατί οι εκλεγμένοι, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες δεν θα είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί η τραπεζική καιροσκοπία θα εκφεύγει από κάθε έλεγχο. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αργά ή γρήγορα. Το καθεστώς, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η αποστολή της. Έχει βέβαια το ρόλο της νομισματικής πολιτικής. Αλλά αυτή η νομισματική πολιτική μέχρι στιγμή έχει λειτουργήσει μόνο προ όφελο των τραπεζών και όχι προ όφελο των κρατών για να αντιμετωπίσει την ένδια και την απασχόληση. Την ανεργία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία θέση από κοινού των ε, χρεών των χωρών και η κάθε χώρα προσπαθεί να διασώσει μόνη τις τραπεζές της και υποφέρουν οι πολίτες λόγω αυτού. Αν μας εμποδίζουν οι συνθήκες, γιατί δεν προχωρούμε σε ένα νέο σύστημα παράλληλο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια δημόσια τράπεζα η οποία θα ασχολείται με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, με την ευρωπαϊκή συνεργασία, με νέα σχέδια ε, επενδύσεων για μια οικολογική μεταστροφή τη οικονομία. Αναφέρατε ακροθυγός κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου το εγχείρημα αυτό της ε, συμφωνίας αυτής για την ε, ανταγωνιστικότητα, δηλαδή περισσότερα χρήματα για τις χώρες οι οποίες ακολουθούν το δρόμο της καταστροφής των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού συμβουλίου. Δεν έχουμε αρκετά περιοριστικά σχέδια, το 2-pack, το 6-pack, το δημοσιονομικό σύμφωνο, ήδη που έχουμε αποφασίσει. Αλλά ποτέ δεν μιλάμε για αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι η Ευρώπη. Μια ανθρώπινη, μια κοινωνική Ευρώπη. Αυτή η ανθρώπινη Ευρώπη θα μας επιτρέψει μονάχα να επιτύχουμε μια δημοκρατική Ευρώπη και να βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ. Για τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Κλέσ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, πρόκειται για την 25η συνάντηση του Συμβουλίου για την οικονομική κρίση. 25 συνέδρια πριν ε, ξεκίνησε μια συζήτηση η οποία δεν μπήκε ποτέ στην ουσία για την έννοια της αλληλεγγύης και την ελαστικότητα που χαρακτηρίζει τον όρο αυτό. Πολλά λέμε για την αλληλεγγύη, κανένας όμως δεν διευκρινίζει περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για μια αλήθεια χωρίς τέλος. Σαν φλαμανδός Αναγνωρίζετε αυτά τα οποία λέω κύριε Πρόεδρο του Συμβουλίου. Ξέρετε για τις μεγάλες οικονομικές ροές, χρηματοδοτικές ροές από την Φλάνδρα στην Βαλονία και από ό,τι θέλετε τώρα να φτιάξετε φαίνεται είναι μια Ευρώπη τύπου Βελγίου όπου οι βόρειες χώρες θα πρέπει να στηρίζουν τις φτωχές νότιες. Δηλαδή θέλετε να βελγοποιήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι αλληλεγγύη είναι αυτή λοιπόν, ποια είναι τα όρια της, ποια η ελαστικότητά της. Ένα άλλο θέμα, ε, τα, η δημοκρατική νομιμότητα των μέτρων που μόλις ανακοινώσατε. Στα συμπεράσματά σας, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, εγώ διαβλέπω κάτι το επαναστατικό. Πώς θα συμμετέχουν ε, τα ε, κοινοβούλια των κρατών μελών σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι επαναστατικό είναι η διατύπωσή σας. Θέτει ερωτήσεις, δεν δίνει απαντήσεις. Τι είδους δημοκρατικός έλεγχος είναι αυτός τον οποίο φαντάζεστε στο μέλλον εφόσον η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση ε, εντάσσεται πλήρως στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Τώρα όσο για την τραπεζική ένωση αυτό θα πρέπει να είναι κάτι φρικτό έτσι όπως το ορίζετε για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Πώς θα μπορέσετε εσείς να δώσετε εγγυήσει στους αποταμιευτές και πώς οι τράπεζες θα είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα κύριε Μπερόζο, είστε εντελώς αδύναμος κύριε Βαν Ρόμπαϊ και γι' αυτό η 25η συνάντησή σας δεν απέδωσε ως συνήθως τίποτα. Uh, Ο κύριος Μπαρόζο, νομίζω στην πρώτη μου εισήγηση μου αρκετά αντικειμενικός και δίκαιος το πώς ε, αποτίμησα το, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όντω, κατέστη δυνατόν να υπάρξει μια σημαντική απόφαση. Βεβαίω, λογικώ οδηγηθήκαμε εκεί από όσα συζήτησαν οι Υπουργοί Οικονομικών. Όμω το γεγονό ότι επίκειτο την επομένη σύνοδο του Συμβουλίου, αυτό βοήθησε του Υπουργού Οικονομικών να καταλήξουν σε αυτή τη σοβαρή απόφαση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Τραπεζική Ένωση δεν είναι απλώς ένα βήμα, ούτε ο εποπτικός μηχανισμός. Ίσως είναι από, τα σημαντικό, από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για τους επενδυτές μας και όσους μας κρίνουν. Εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Σεπτέμβριο έχει κάνει πρόταση επίσημα, αλλά και προηγουμένως προσπαθήσαμε. Εάν θυμάστε, εγώ ε, είχα ζητήσει από τα κράτη-μέλη και στο παρελθόν να τα συζητήσουν αυτά. Υπήρξε απορριπτική στάση, μόνο και μόνο γιατί περάσαμε από τον μηχανισμό του EBA και οι εθνικοί επόπτες ε, τελικά υπερίσχυσαν. Το ψήφισε και το κοινοβούλιο με συναπόφαση. Όμως, αυτό που δεν ήταν εφικτό το 2008-2009, να βλέπουμε ότι κατέστη πλέον δυνατό το 2012. Οπότε μπορούμε να λέμε λογικώς ότι ε, κάποια ενδεχόμενα είναι ακόμη ανοιχτά. Τι εννοούμε όμως με αυτό. Υπάρχουν ε, συζητήσει με το, στα επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πάει παραπέρα. Η τέταρτη έκθεση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το ίδιο. Αλλά να καταλαβαίνουμε και το εξής. Δεν αγγίζουμε την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Όταν μιλάμε για συντονισμό, εξάντε, για τους εθνικούς προπολογισμού, πρέπει να κατανοούμε ότι αυτό είναι πρόκληση και είναι κάτι που προκαλεί εντάσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Το ίδιο και η δημοκρατική λογοδοσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν, είναι και θα είναι, ελπίζω και στο μέλλον, ε, σταθερή στο ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις εθνικές δημοκρατίες με την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η βάση για, τις ευρωπαϊκές, για την ευρωπαϊκή δημοκρατία είστε εσεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε άμεσα εκλεγμένοι από του πολίτε και είστε επιφορτισμένοι με την ευρωπαϊκή κυριαρχία, όπως είπε και ο κύριος Σαλόμ. Όμως, όταν μιλάμε για εθνικούς προπολογισμού, είναι φυσικό και τα εθνικά κοινοβούλια να θέλουν να συμμετάσχουν στις όλες τις διαπραγματεύσεις. Οπότε, όχι μόνο χαίρομαι για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και κάποιε συζητήσει που είχα στο περιθώριο πρέπει να πω ότι ήταν ικανοποιητικέ. Γιατί κάποιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μα είπαν: Ήταν ενδιαφέρουσε οι ιδέε σα, αλλά δώστε μα και λίγο χρόνο να τα σκεφτούμε. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αίσθηση ότι έχουμε περάσει στα ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα και γι' αυτό πρέπει να γίνει συζήτηση ευρωπαϊκού επίπεδου. Όταν σα συνάντησα πριν το Στρασβούργο, σα μίλησα και για τι ε, επόμενε ευρωεκλογέ. Είπα ότι θα είναι μια καθοριστική στιγμή για να γίνει πολιτικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το είπε και η κυρία Χάρμ. Η πραγματικότητα ω τώρα ήταν η εξή. Οι ευρωεκλογέ ήταν μια συλλογή από 27 εθνικές εκλογές. Ας έχουμε για μια φορά μια πραγματική συζήτηση, ευρωπαϊκής εμβέλειας, με ψηφοφόρους, με πλατφόρμες συζήτησης, με πραγματική συμμετοχή, ώστε όλες οι φιλευρωπαϊκές δυνάμεις να προβληθούν και να εξηγήσουν στι χώρε του, όχι μόνο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, στι πατρίδε του, ποιε είναι οι διαφορετικέ επιλογέ, ποια είναι τα ενδεχόμενα. Νομίζω αυτό είναι ο μόνο τρόπο. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει στα πραγματικά ευαίσθητα ζητήματα για όλου. Και από αυτή τη σκοπιά καλά κάναμε και προχωρήσαμε με την Τραπεζική Ένωση και τον ενίο εποπτικό μηχανισμό και τη δέσμευση των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων για την ταχεία έγκριση τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρόκειται να δημοσιευτεί τώρα για τον ενιαίο μηχανισμό αντιμετώπιση. αλλά και το άνοιγμα για τον εξάντε συντονισμό των εθνικών πολιτικών ήταν θετικό. Όλα αυτά για μένα ήταν θετικά. Αλλά σίγουρα υπάρχουν διαφορέ μεταξύ του δικού μα αποτυπώματο και τη τέταρτη έκθεση τη Προεδρία. Δεν ήταν όλοι όμω έτοιμοι να τα εγκρίνουν ε, εξ ολοκλήρου σε αυτό το Συμβούλιο. Είναι σαφές αυτό. Αλλά τι ευκαιρία τον μπροστά μας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία να ξεκινήσει η όλη συζήτηση, διότι πιστεύω επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, δεν έχουμε ξεφύγει από την κρίση. Είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι ξεφύγαμε. Ειδικά αν σκεφτούμε την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στι διάφορε χώρε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά ακόμη και στη διακυβέρνηση τη ε, Νομισματική Ένωση έχουμε ακόμα πολλή δουλειά η καλύτερη, η κατάσταση είναι τώρα λίγο καλύτερη πριν, σε σχέση με πριν από λίγο καιρό. Όχι επειδή πήραμε μια-δυο αποφάσεις, αλλά υπάρχει πλέον μια δυο αποφάσει. αλλα υπαρχει απόκριση. Και κάποιε μεταρρυθμίσει προχωρούν σε κάποια κάτι Δηλαδή τα δημοσιονομικά διορθώνονται, το έλλειμμα ακολουθεί πτωτική πορεία είναι πολύ σημαντικό ότι μιλήσαμε για τον ε, επιποπτικό μηχανισμό. Αυτό το αντιμετώπισαν πολύ θετικά οι επενδυτέ. Το άκουσαν με ευνοϊκό αυτοί. Και μην ξεχνάτε ότι αποφύγαμε και την πτώχευση στην Ελλάδα. Πολλοί αναλυτέ, πολλοί οικονομολόγοι προέβλεπαν πτώχευση τη Ελλάδα πέρσι. Τώρα φτάσαμε στο τέλο τη φετινή χρονιά και η Ελλάδα δεν ε, έφτασε σε αυτή την κατάσταση μπορούμε να στηρίξουμε το ευρώ, στηρίζουμε την νομισματική ένωση και αυτό είναι μια διαδικασία δυναμική. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν και μαζί με τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ΕΝΤΗ βλέπουμε ότι καταφέρνουμε να διασφαλίσουμε την οικονομική και νομισματική ένωση και να την εμβαθύνουμε. Γι' αυτό πρέπει να, να συνεχίσουμε με αυτή την πυγμή ε, και την αποφασιστικότητα η αυτοπεποίθηση χάνεται πολύ εύκολα σε μια στιγμή, αλλά δύσκολα να κτάτε. Θέλει χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα χρειαστεί χρόνο για να υπάρξει ξανά πίστη στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι θετικό να υπάρχουν ανοιχτά ενδεχόμενα. Και η φιλόδοξη απόκριση που θα έχουμε είναι αυτή για την οποία πολεμάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ισχυρότερη νομισματική ένωση σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχω περισσότερα να προσθέσω σε αυτά τα οποία μόλις είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Κάποιες όμως συμπληρωματικέ παρατηρήσεις. Ήδη από τον μήνα Ιούνιο, όταν καταθέσαμε την πρώτη μας έκθεση, είχαμε μιλήσει για τέσσερους βασικούς τομείς, τέσσερους building blocks, λέει στα αγγλικά ο Πρόεδρος έχουν επίθετα και ονόματα που δεν καλύπτουν πλήρως τα παιδεία, ε, πολιτική, οικονομική, νομισματική ένωση κτλ. Από, τον, από τις 13 Ιουνίου και μετά δηλαδή συνεργαστήκαμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Δεν ε, ζητήσαμε το Συμβούλιο να εγκρίνει τις προτάσεις της Επιτροπής όσοι είχαν τότε. Εμείς είχαμε ανοίξει μια τέτοια μακροπρόθεσμη προοπτική και ε, σιγά σιγά βαθμιαία στα πλαίσια αυτής της σταδιακής αντίληψης που εξέθεσα προτείναμε για κάθε ένα από αυτούς τους βασικούς τομείς να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν την ίδια κατεύθυνση και τον ίδιο προσανατολισμό. Χαράξαμε δηλαδή μία μακροπρόθεσμη πολιτική και ε, χαράξαμε τα κεφάλαια με τα οποία θα ασχοληθεί ή ασχολήθηκαν τα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούστηκαν για την Πιστοτική Ένωση, για την Τραπεζική Ένωση. Υπήρξαν πολύ σημαντικά βήματα εκεί και τα βήματα αυτά έγιναν σε επίπεδο 27 χωρών. Όλα τα μέλη δηλαδή του Συμβουλίου πήραν μέρος πήραν μέρος στη λήψη των αποφάσεων ακόμα και ε, με τις χώρες που είπαν ότι δεν θέλουμε να πάρουμε μέρος στην Τραπεζική Ένωση και στο σύστημα εποπτείας. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θα συμφωνήσουμε. Ναι κύριε Ντόλ και η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον, συμφώνησε να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία με 27 υπογραφές. Ένα δεύτερο θέμα στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης καταλήξαμε σε μία λήψη θα έλεγα απόφασης επί της αρχής για τον μηχανισμό επίλυσης κρίσεων και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προτείνει σε εύθετο χρόνο και μάλιστα κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για τον χρονισμό. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με την ενιαία μορφή εποπτείας. Τον Ιούνιο λοιπόν είχαμε πάρει μια απόφαση επί της αρχής και προσπαθήσαμε να εξελίξουμε την απόφαση αυτή. Χαιρετίζω εδώ τις προσπάθειες των Υπουργών Οικονομικών, αλλά μην φανταστείτε ούτε και μία στιγμή, ακόμα και αν το Συμβούλιο είχε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει μία απόφαση πριν από τον μήνα Δεκέμβριο, ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτή την απόφαση. Τον Οκτώβριο είχαμε πει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ισότιμα και οι χώρες που είναι εκτός ζώνης ευρώ. Και είχαμε πει επίσης ότι θα θέλαμε να αλλάξει και η διαδικασία ψηφοφορίας στην αρχή την τραπεζική έτσι ώστε να μην αποκλειστεί καθνής και να παραμείνει η τραπεζική αγορά μια ενιαία αγορά. Αν δεν είχε υπάρξει λοιπόν η απόφαση αυτή δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Τώρα για τη Δημοσιονομική Ένωση. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να καταλήξει σε μια συμφωνία για το λεγόμενο διπλό πακέτο. Είναι απαραίτητο συστατικό αυτής της μορφής της Ένωσης. Μετά από αυτά τα οποία κάναμε και με το εξαπλό πακέτο, όπως επίσης και με την Δημοσιονομική Συμφωνία, Νομίζω ότι το διπλό αυτό πακέτο, το 2 είναι ένα σημαντικό βήμα. Έχουν ήδη συντελεστεί βήματα πρόοδου. Έχουμε προχωρήσει στην Οικονομική Ένωση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα, ακόμα και εκεί. Ε, θα έλεγα ότι δεν είμαστε βέβαια σίγουροι ότι οι χώρες θα ακολουθήσουν τις συστάσεις αυτές, ακόμα και αν είναι συστάσεις οι οποίες είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Από την άλλη, έχουμε το σύστημα των μακροοικονομικών ανισορροπιών και εδώ δημιουργούμε ένα τέτοιο μέσο το οποίο προτείνεται στα πλαίσια του εξαπλού πακέτου. Ίσως όμως να υπάρξουν καθυστερήσεις. Για να προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα και για να εμπλακούν όλες οι χώρες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όλες οι χώρες έχουν ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις θα πρέπει να αναλυφθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και οι συμβάσεις αυτές, τα σύμφωνα αυτά, είναι κάτι που σέβεται με τις εθνικές αρμοδιότητες πλήρως, αλλά αυτές οι συμβατικές υποχρεώσεις που είναι καρπός διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζουν την κάθε χώρα για να προχωρήσει ταχύτατα και ακόμα περισσότερο στον δρόμο της σύγκλησης της πολιτικής και οικονομικής. Δεν είναι πειθαρχικά συμβόλαια αυτά, είναι συμβόλαια, είναι σύμφωνα που έχουν σαν στόχο την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την απασχόληση. Είναι μια έννοια πλούσια και πολλαπλή. Δεν πρόκειται για κυρωτικές αποφάσεις και συμβάσεις, πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες έχουν θετική, θα έλεγα, θετικό περιεχόμενο. Σεβόμεθα πλήρως τις εθνικές αρμοδιότητες και ταυτόχρονα υποχρεώνουμε την χώρα να προχωρήσει στα πλαίσια των καθορισμένων στόχων Τη στρατηγικής Ευρώπη 2020. Για τον δημοκρατικό έλεγχο θα πρέπει να ξεκινήσουμε οργανώνοντας τον έλεγχο αυτό στους τομείς τους οποίους είναι απαραίτητος και δεν θα πρέπει εμείς να μπλέξουμε σαν Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια των Κραντών Μελών. Αυτή είναι δική σας δουλειά και δεν θα δώσουμε οδηγίες εμείς. Πάντως βασική αρχή είναι ότι δημοκρατικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων του καθενός. Να πω λοιπόν ότι αυτό το Συμβούλιο είναι ένα νέο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Στην εκτέλεση ενός μακροπνού και μακροπόθεσμου σχεδίου. Προφανώς έχουμε εστιάσει περισσότερο στο Βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αυτά τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα στους επόμενους 6 μήνες. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές όμως οι οποίες θα υλοποιηθούν δεν θα κρατήσουν για 6 μήνες, ελπίζω για 60 χρόνια. Όταν συμφωνήσουμε για ένα μηχανισμό εποπτείας δεν είναι για το βραχυπρόθεσμο μονάχα μέλλον. Ο μηχανισμός επίλυσης δεν είναι μονάχα για τους επόμενους 6 μήνες. Θα εργαστούμε για 6 μήνες ίσως, αλλά εννέα μήνες για τη φύση είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονική περίοδος. Από μέσα εννέα μήνες η μη ζωή γίνεται ζωή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έξι μήνες είναι αρκετοί όμως, είναι πολύ οι έξι μήνες. Δεν ξεπερνάμε τα φυσικά όρια. Υπάρχουν κάποιες ιδέες οι οποίες δεν έχουν οριμάσει ακόμα, θα πρέπει να εργαστούμε, όπως είπε και ο πρόεδρος Κομισιόν. Αυτό το οποίο ήταν αδύνατον ή ανέφικτο πριν από τρία χρόνια είναι τώρα δυνατό φτάνουμε τώρα σε κάποιους σκληρούς πυρήνες κυριαρχίας, αλλά και σε κάποιους σκληρούς πυρήνες σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να το πούμε. Μπαίνουμε τώρα σε τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα, αλλά πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν υπάρχει πια η πίεση των αγορών, θα πρέπει να υπάρξει πίεση των θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό η έκθεση αυτή, οι εκθέσεις αυτές που εκδίδουμε είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί εξακολουθούν να διατηρούν την πίεση των θεσμικών οργάνων. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα. Αλλά δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να γίνουν από την πρώτη στιγμή. Αλλά είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την κατεύθυνσή μας. Για αυτούς οι οποίοι κάνουν συγκρίσεις με τον Άγιο Βασίλη ή με ορισμένους άλλους, με τους άγγελους, τους ευχαριστώ. Αλλά ότι με συγκρίνουν με αγγέλους, ίσως δεν έχουν δίκιο, δεν είμαι ούτε άγγελος ούτε διάβολος σε αυτά τα θέματα. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε απόλυτη υπεπίγνωση του γεγονότος ότι είναι μακρός, μα, μακρύς ο δρόμος, ότι κάποιες από τις χώρες μας περνάνε μια χρονική περίοδο μεγάλες δυσκολίες. με τον πληθυσμό τους και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός τους, τους ε, βοηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο με το μηχανισμό αυτό αλληλεγγύης και έχουμε απόλυτη επίγνωση των προβλημάτων και όσων παραμένουν να γίνουν. Αλλά για ε, τούτων λεχθέντων ήταν μια θετική εβδομάδα για την Ευρώπη και έχουμε προχωρήσει στον δρόμο στον οποίο θέλουμε να κινηθούμε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω να ευχηθώ σε όλους σας καλές γιορτές, καλή, καλό νέο έτος και καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο χρόνο λέει και στα φλαμαντικά ο κύριος Φανρομπάη. Υπάρχουν οι άγγελοι οι οποίοι ενούν τον Κύριο στον ουρανό και λένε καλά Χριστούγεννα και αυτοί. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εννέα μήνες κύριε Φων Ρομπάι. Επιτρέπω στον εαυτό μου να σας πω ότι στην αρχή αυτής της περίοδου εννέα μηνών λαμβάνει συνήθως κάποιο γεγονός το οποίο είναι πιο ευχάριστο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ίδιο. Αυτό νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητο. Δίνω τώρα το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Κλάς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το δημοκρατικό έλλειμμα, κύριε Μπαρόσο και κύριε Βαν Ρομπάη, επιλέξατε να απαντήσετε με πάρα πολύ ε, θολά λόγια θα έλεγα. Γενικά δεν δώσατε απαντήσεις. Ίσως το κάνατε για να μην προκαλέσετε το κοινοβούλιο. Αλλά αν θέλετε όμως η κοινή γνώμη να ενδιαφερθεί και αν ε, πραγματικά δεν θέλετε να απομακρυνθούμε από την πραγματικότητα θα πρέπει δυστυχώς να αλλάξετε τις θέσεις σας. Ο κύριος Λογιαρίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπαρόσο λέγοντας ότι δεν βγήκαμε από την κρίση Είπατε όμως πρόεδρε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς αυτό για τους πληθυσμούς που υποφέρουν. Αναφερθήκατε στην Ελλάδα η κατάσταση και στην Πορτογαλία, την Ισπανία και στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι πολύ δύσκολη για τους πληθυσμούς. Εκπλήσωμε που δεν το συζητάμε αυτό. Εκπλήσωμε που δεν θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις γύρω από την αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις πιθανότητες αναπροσανατολισμού. Λυπάμαι που δεν μιλάμε για τα χίλια δις φορο, ε, ε, φοροδιαφυγής που σημειώνονται στο εσωτερικό της Ευρωζώνης που θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε για την δημιουργία των ταμείων που θα στηρίξουν τις τράπεζες απευθείας και όχι μέσω των κρατών και τα χρήματα τα υπόλοιπα να χρησιμοποιηθούν για την κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια δεν απαντάτε. Μιλάτε για οικονομική ε, και κοινωνική διάσταση. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει ένα κοινωνικό σύμφωνο. Ευχαριστώ κύριο Χέλμερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρόσο και τον κύριο Φαρομπάι για τις απαντήσεις που μου δώσανε. Αλλά οι απαντήσεις δείχνουν πιο σαφώς από ότι θα μπορούσα να το κάνω ο ίδιος εγώ ότι έχουν κάτι να πούν αλλά δεν είναι απάντηση αυτό. Ο κύριος Μπαρόσο χαίρεται για το γεγονός ότι υποστηρίξαμε το ευρώ. Θα ήταν καλύτερα να υποστηρίξετε τους πολίτες οι οποίοι έχουν βασανιστεί στον ε, βωμό του ευρώ. Μιλάτε για περισσότερη δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά η δημοκρατία απαιτεί ένα Δήμο, απαιτεί μια κοινή γνώμη που να είναι πανευρωπαϊκή και αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μια δημοκρατική Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μονάχα σαν Ευρώπη δημοκρατικών κρατών μελών η δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια φάσα, δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Ακούσαμε να μιλάτε για πιο πολύ δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση. Μα μέσα σε μια ενιαία οικονομική ζώνη έχετε εγκαταλείψει τους μοχλούς της νομισματικής πολιτικής. Ίσως χρειάζεται ακόμα περισσότερη διαφορά στις δημοσιονομικές πολιτικές για να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό στην Ευρωζώνη. Είδαμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες Καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν έχει επιτύχει. Θέλαμε περισσότερη εμπιστοσύνη, θέλαμε εργα... θέσεις εργασίας, ε, ανάπτυξη, τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε πετύχει. Και εσείς κύριε Φαν Ρομπάι είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο με βρίσκει σύμφωνο, είπατε ότι η Ευρώπη θα επιβιώσει μονάχα αν είναι ανταγωνιστική. Μα τι κάνετε για να την κάνει την Ευρώπη ανταγωνιστική. Υπάρχει ένα τεράστιο βάρο υπερβολική ρύθμιση, το οποίο πρέπει να το ξεφορτωθούμε αν οι Ευρωπαϊκέ οικονομίε θα ξαναγίνουν ανταγωνιστικέ. Χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους και χρειαζόμαστε κυρίως να σταματήσουμε αυτές τις παράλογες πράσινες πολιτικές της Ευρώπης που οδηγούν στην πιο ακριβή ενέργεια στον κόσμο. Δεν θα μπορέσουμε με αυτές τις τιμές ενέργειας να είμαστε ποτέ ανταγωνιστικοί. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα να προσφέρετε. Το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει πια η εποχή του. Το ευρώ θα πρέπει να του δοθεί μία μορφή ευθανασίας πια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο με την ε, διάσκεψη κορυφή όσο έλαβε χώρα. Και απλώ έχω να κάνω μια παρατήρηση για τον κύριο Ντόλ, αν με ακούει. Ίσως θα πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα οποία κηρύττει. Γιατί μιλάτε για ένα πολιτέ πλαίσιο και μετά αρχίζετε να επιτίθεστε κατά της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά και η Ολλανδία και η Γερμανίδα καγκελάριο δεν συμφωνούμε με την πρότασή να αυξηθεί ο προπολογισμό κατά 5%. Αν προσπαθείτε να βρείτε ένοχου για τη μη συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξεκινήσετε με τη δική σα πολιτική οικογένεια. Και ίσω και ο κύριο Μπαρόσο θα πρέπει να εξετάσει τι γίνεται, που είναι δική του πολιτική οικογένεια. Δεν είμαστε λοιπόν μόνο εμεί οι συντηρητικοί. Ο λόγος για τον οποίο τα είπατε όλα αυτά είναι γιατί δεν έχετε επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Προσπαθήστε να εξηγήσετε στους, πραγματικ... στους απλούς πολίτες ότι εσείς χρειάζεστε περισσότερα λεφτά και αυτοί πρέπει να κάνουν οικονομίες. Κυρία Χάρμς. Θα ήθελα να επανέλθω στο ρόλο του κυρίου Ντράγκη. Κατά τη δική μου άποψη, ο κύριος Ντράγκη παίζει εκτός του θεσμικού πλαισίου. Και επομένως τα χρήματα αυτά τα οποία οδήγησαν στις απεριόριστες νομισματικές συλλαγές του κ. Ντράγκη είχαν εκφύγει πλήρως από οποιοδήποτε δημοκρατικό έλεγχο. Πιστεύω ότι ο ρόλος του κ. Ντράγκη είναι ένας ρόλος ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβουλευτικός ρόλος. Η εμβάθυνση όμως και η οικονομική ολοκλήρωση ε, εναπόκειται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν μπορεί να γίνεται αυτό με δημοκρατικά ελεγχόμενο τρόπο αν επαφίεται μονάχα στον κύριο Ντράκη και να περιμένω από τον κύριο Ντράκη να σώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό έργο είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε εκ των υστέρων να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, όταν δίνονται από τη μια μεριά υποσχέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα στον πληθυσμό. Αυτό λοιπόν είναι μια παράληψη την οποία δεν μπορούμε να την ε, αποδεχόμαστε πια. Κύριο Φεχόφστατ, χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Όταν μιλούσαμε για τους εννέα μήνες, ε, ίσως είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά το σημείο της σύλληψης εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί πράγματι θα έπρεπε να υπάρξει μια τέτοια προσπάθεια έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα θετικό συμβάν, σε ένα καλό συμβάν. Ε, για το πρώτο θέμα, για τις ε, συμβάσεις αυτές ε, και τα σύμφωνα με τα διάφορα κράτη-μέλη. Εμείς διαφωνούμε σαν Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε με τέτοιες συμβάσεις διαφορετικές αναχώρα να προχωρήσουμε σε μια σωστή ενιαία πολιτική όχι συμβάσεις, όχι συμβόλαια. Εμείς δεν είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση που υπογράφει μια συμφωνία και με ένα συμβόλαιο με μια άλλη επιχείρηση. Απαιτείται μια διαφορετική στρατηγική σε όλους τους τομείς τους οποίους αναφερθήκατε. Και τέλος, σχετικά με το διπλό πακέτο. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια νέα πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε ακριβώς πώς θα αντιδράσει στην πρόταση αυτή. Είναι μετριοπαθής, εν πάση περιπτώσει, η πρόταση αυτή. Μπορεί να προέλθει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά κάτι σημαίνει η πρόταση αυτή. Όταν το Συμβούλιο σας ζητά να κάνετε ένα εποπτικό μηχανισμό, το κάνετε. Και καλά κάνετε. Όταν το Συμβούλιο σας ζητάει να κάνετε μια πρόταση για μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ε, θα το κάνετε. Είναι συμβατός όμως ο μηχανισμός αυτός για όλες τις τράπεζες με τις συνθήκες. Αν είναι κάτι τέτοιο, ε, τότε ίσως να μην είναι τόσο ε, συμβατό το Ταμείο για την απόσβεση των χρεών. Κύριος Κεραίρο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προηγουμένως έλεγα ότι ήταν κάπως άτομη η προσέγγιση σε σχέση με την ανάπτυξη όταν όλα αφορούσαν την ε, εδραίωση των δημοσιονομικών. Από τη μία πλευρά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μιλάνε για πολιτικές περιεκτικές και αηφόρες. Αλλά με τη βάση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συζήτηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι προγνώσεις σε ό,τι αφορούν την ε, δημοσιονομική εδραίωση ήταν λαθασμένες. Δεν έχει εκτιμηθεί σωστά ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής. Ο κύριος Ρεν έχει προτείνει ήδη στη Σοσιαλιστική Ομάδα να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ οικονομολόγων τη Κομισιόν και εξωτερικών οικονομολόγων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλύτερη μεθοδολογική συμφωνία σε σχέση με την εκτίμηση των Τι Θεωρούμε ότι είναι θετικέ οι διαφοροποιημένε δημοσιονομικέ πολιτικέ για την ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη για το 2013. Τόνισα λοιπόν ότι είναι θετικό το ότι γίνεται κάποια μνήμα κοινωνικό τομέα αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η δική μου πολιτική ομάδα δεν θέλουν κοινωνικές μνήες στα άλλα τέσσερα μπλοκ. Θέλουν ένα ιδιαίτερο μπλοκ το οποίο αφορά τα κοινωνικά θέματα, τον κοινωνικό πυλώνα. Ένα μπλοκ λοιπόν το οποίο θα είναι και στεναρό και υποχρεωτικό και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊ... το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σύμφωνο που θα έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίσης όπως είπε και ο κύριος Φαν η σχέση μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ο, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα και αν δεν αλλάξουμε τίποτα και αφήσουμε κατά μέρο τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εμεί έχουμε την απέτηση όλα τα θέματα τη οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια συναπόφαση με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερο αυτό θα πρέπει να είναι υπόλογος εναντί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιμένουμε ότι οι τρόικες με τις διάφορες εκφάνσεις τους πάλι θα πρέπει να είναι υπόλογοι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μπαρόσο μίλησε για επίπεδο φιλοδοξίας. Είναι σωστό να πούμε ότι η μεγαλύτερη φιλοδοξία βρίσκεται στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι η Κομισιόν είναι πιο φιλόδοξη από ότι δεν είναι, ότι, θα λέ, όταν δεν έλεγα ότι η Κομισιόν είναι πιο φιλόδοξη από τον πρόεδρο Συμβουλίου και ο πρόεδρο του Συμβουλίου πιο φιλόδοξο από τα κράτη-μέλη. Αν όμω θέλουμε τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, ο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή είναι πάντα μηδέν. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει πραγματικά κοινή εργασία σε όλα αυτά τα θέματα. Και επειδή είμαστε κοντά στι γιορτέ των Χριστουγέννων και όπω όλοι έχουν κάνει ευχέ, ίσω ελπίζουμε ότι σε 9 μήνε θα προκύψει κάτι διαφορετικό, το οποίο θα κάνει δυνατό να υπάρξει ένα ταμείο από κοινού ε, του χρέους και αυτοί οι οποίοι είναι θρησκευόμενοι θέλω να τους υπενθυμίσω ότι, ότι μέχρι ότου ο, ότι ο Πάπας μπορεί να αποφάσισε ότι δεν είναι απαραίτητα τα βόδια στη φάτνη αλλά οι άγγελοι είναι πάντα απαραίτητοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρε Βαν Ρομπάι θα πρέπει να σας συγχαρούμε γιατί καταφέρατε να εγγράψετε την πολιτική της ασφάλειας και της άμυνας στην ημερήσια διάταξη. Καιρός ήταν εδώ και τρία χρόνια αυτή η νέα μείζων αυμοδιότητα μας ανήκει και δυστυχώς διαβάζοντας βέβαια τα συμπεράσματα δεν υπάρχει κάτι εκεί, δεν, υπάρξει, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αναφορά στις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ, στην εξωτερική πολιτική, ε, στη μόνιμη διαφθορτμένη συνεργασία. Ε, γενικά δεν υπήρξε αναφορά στα θέματα άμυνας ε, και δεν υπήρξε θέμα καν συζήτησης για την κοινή ανάλυση μιας μορφής απειλής. Εμείς θα πρέπει να δούμε τι έχουμε να κάνουμε γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις στους τομείς αυτού σήμερα. Επί της ουσίας τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία αφήσετε σε εκκρεμότητα. Μετά από τρία χρόνια κρίσης μπορέσαμε να απαντήσουμε σε ένα πρόβλημα ποιος είναι ο τελευταίος τελικός αποφασιστικός δανειστής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν με τους όρους που όλοι τώρα πλέον καλά γνωρίζουμε. Από την άλλη το Συμβούλιο δεν έχει θέσει την εξή ερώτηση, πιο δύσκολη, ποιος θα είναι ο, ο, ο, φορολο, ο, ο πολίτης ο οποίος φορολογείται που θα είναι ο τελευταίος ο οποίος θα δώσει τα χρήματα. Αυτή είναι μια συζήτηση πολιτική και σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τους ιδίους πόρους και τις ίδιες ανάγκες της ζώνης ευρώ. Η συζήτηση αυτή για τη δημοσιονομική ικανότητα, αν θέλετε, της Ένωσης δυστυχώς χάθηκε. Με την ελάφρυνση του χρέους ε, με την ελάφρυνση του χρέους ε, της Ελλάδας, ε, με τις πιστοτικές νέες μορφές εποπτείας, με τις, αυτές τις συμφωνίες, συμβόλαια με τα κράτη-μέλη, είναι σαφές ότι οι φορολογούμενοι θα χρειαστεί να πληρώσουν. Ποιοι φορολογούμενοι και πότε και πόσο. Τίθεται λοιπόν το θέμα αυτό και είναι πολύ δύσκολο. Όταν πρόκειται για να συντονίσουμε πολιτικές οι οποίες είναι πάντα εθνικές αρμοδιότητες και το θέτει το πρόβλημα αυτό κύριος Μπαρόσο, ποιος θα πρέπει να είναι ο, αυτός που παίρνει την απόφαση σε τελική φάση, σε αποφασιστική φάση. Το σύστημα αυτό του Συμβουλίου παρουσιάζει κάποια όρια. Σε περίοδο κρίσης βέβαια είναι σαφές ότι είναι νόμιμο η απόφαση να λαμβάνεται εκεί. Αυτή τη στιγμή όμως κατασβεστεί η πυρκαγιά, μετατρέπεται ένα τέτοιο συμβούλιο σε διπλωματική διάσκεψη. 27 εθνικές πραγματικότητες δεν συνιστούν, αν θέλετε, μια τέτοια μορφή όπως απαιτείται σήμερα κάποιες αποφάσεις απαιτείται να υπάρξει κοινοβουλευτική έγκριση όπως για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Αλλά αλλιώς φοβάμαι ότι γίνονται συζητήσεις και προτάσεις τις οποίες θα ξεχνάσουμε αμέσως. Το τελευταίο συμβούλιο που είχε σαν στόχο την ανταγωνιστικότητα δεν αναφέρθηκε καθόλου ούτε στην Ατζέντα 2020 ούτε στο Σύμφωνο Ανάπτυξης είχαν εδώ και έξι μήνες πει ότι θα δώσουν 120 επιπλέον δις και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να πληρώσει και να κλείσει τους λογαριασμούς του 12. Λοιπόν, ε, τι νόημα έχει λοιπόν να λέμε μεγάλα λόγια αν δεν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε αυτά. Το Συμβούλιο έχει δίκιο που θέτει ερωτηματικά για τον κοινοβουλευτικό και διακοινοβουλευτικό έλεγχο της ίδιας του της δράσης και δραστηριότητας. Θα πρέπει να θέσει ερωτήσεις όμως και για τον τρόπο που λειτουργεί. Ε, δεν πρόκειται για ένα συλλογικό όργανο ε, των ε, ηγετών των κρατών μελών όπως το παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα μόνιμο ε, φόρουμ όπου θα συνεδριάζει ένα αντίστοιχο του G20. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τόσο ζωντανή αυτή ανταλλαγή απόψεων. Θα ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν η τελευταία συνέλευση των Προέδρων του 2012 και βέβαια ήταν ανοιχτή σε όλους τους ε, βουλευτές. Η επόμενη συνέλευση των Προέδρων λαμβάνει χώρο, χώρα στις 10 Ιανουαρίου και σας εύχομαι να κατέβουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια αγγέλων οι οποίοι θα συμβάλλουν σε ένα ευτυχισμένο αλλά και υγιές 2013 και από τη δική μου πλευρά ελπίζω ότι θα μπορέσει το 2013 η ειρήνη που έχουμε στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει και ειρήνη και σε άλλες υπήρους του κόσμου που δοκιμάζονται σήμερα. Σας εύχομαι λοιπόν ε, χρόνια πολλά και κλείνω τη συνεδρίαση.